Benvenuti a tutti, diamo inizio alla Λοιπόν, ξεκινάμε. Παρακαλώ, καθίστε. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρείται δεκτή η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα εδώ να σας πληροφορήσω ότι υπάρχει διερμηνία, αν δεν κάνουμε λάθος, σε όλες τις γλώσσες και ευχαριστώ την επιμελητία. Λοιπόν, πέραν της έγκρισης των πρακτικών, δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, αν υπάρξουν μέχρι το τέλος ε, της ε, συνεδρίασης θα συμπληρωθούν, αλλιώς θεωρούνται δεκτά ως έχουν. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ο συνήθως ότι η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο web streaming του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον Σουηδό Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Έσκιλ Έρλαντσον. Για μια ακόμη φορά είναι παρόν στις εργασίες μας και δίδω το λόγο αμέσως στον κύριο Υπουργό για να μας κάνει τον απολογισμό της Σουηδικής Προεδρίας που χαρακτηρίζεται και από τη θέση σε ισχύ φυσικά της συνθήκης της Λισαβόνας όπως επίσης και την εκκίνηση της διαδικασίας συναπόφασης για την Γεωργία. Εσκυλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πάολο, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Σχεδόν έχει περάσει ολόκληρος μήνας που παρέδωσα τη σκητάλη στον Ισπανό συνάδελφό μου. Ήταν συναρπαστικό και ενδιαφέρον το εξάμεινο της Σουηδικής Προεδρίας. Είχαμε πολύ ε, αξιόλογα επιτεύγματα δεδομένης της ε, σύντομης διάρκειας της Προεδρίας. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε ε, το περασμένο φθινόπωρο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος ε, και ευχαριστημένος ε, για τις επιδόσεις μας. Η θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας συνεπάγεται μεγάλες αλλαγές και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο. Μεταξύ των οποίων και αλλαγές στον τομέα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία ούτως ώστε με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να θέσετε επιτυχώς σε εφαρμογή τη νέα συνθήκη. Εν ώψη προεδρία Προεδρίας είχαμε τρεις προτεραιότητες. Ε, το, η βασική ήταν η αλλιευτική πολιτική. Με το τέλος της Προεδρίας είχαμε καταφέρει να εγκρίνουμε 25 νομοθετήματα. Τώρα θα επικεντρωθώ στα θέματα δικού σας ενδιαφέροντος, το, τα τρόφιμα, οι κλιματικές αλλαγές και οι παγκόσμιες προκλήσεις. Η επισητιστική ασφάλεια και η κατοχήρωσή της σε παγκόσμιο επίπεδο είναι βασική προτεραιότητα. 9 δις θα είναι ο πληθυσμός της γης κατά πάσα πιθανότητα το 2050 το Νοέμβριο έγινε σύνοδος κορυφής ε, για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα στα πλαίσια της ε, διάσκεψης του ΦΑΟ και λήφθησαν σοβαρές ε, αποφάσεις. Μεταρρύθμιση της Επιτροπής του ΦΑΟ για την κατοχήρωση επιστήτιστικής ασφάλειας και δρομολόγηση τη παγκόσμια εταιρική σχέση στον τομέα τη γεωργία, του ασφαλού εφοδιασμού σε τρόφιμα και τη διατροφή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον ασφαλή εφοδιασμό σε τρόφιμα και επί Σουηδικής Προεδρίας έγινε διάλογος για την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή των διεθνών στόχων Λοιπόν για επιστημιστική ασφάλεια. Περαιτέρω παγκόσμιε προκλήσει και ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν εντατικά το φθινόπωρο είναι, η σχέση ανάμεσα στη γεωργία και το κλίμα. Αυτό συνιστούσε και δική μου προτεραιότητα επί Σουηδική Προεδρίας. Όπως σας είπα, ε, όταν ήρθα να σας επισκεφθώ το Σεπτέμβριο. Τον Ιούλιο ε, ε, έγινε συζήτηση στο Συμβούλιο επί τη βάση του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμογή της γεωργίας και της ανάπτυξης αγροτικής υπαίθρου στις νέες κλιματικές αλλαγές. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία του ζητήματος και φυσικά θα έχει ε, αυξανόμενη βαρύτητα στο μέλλον. Ε, είμαι πεπισμένος ότι θα αφιερώσουμε σε αυτό το θέμα πολύ χρόνο, δηλαδή να καταφέρουμε να συνδέσουμε τη γεωργία με τις νέες ε, κλιματικές αλλαγές και την πολιτική που θα ακολουθήσει η Ένωση μετά το 2013. Θα εμβαθ... Στη συνέχεια έγινε άτυπο συμβούλιο το Σεπτέμβρη στο Βέξχε και ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό διότι όλοι οι συνάδελφοί μου στο Συμβούλιο ομονόησαν σχετικά με την σημασία της σχέσης ανάμεσα στη γεωργία και το κλίμα και όλοι αναγνώρισαν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών ε, των αερίων του ε, θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ε, στέφθη με επιτυχία το Συμβούλιο αυτό και θα ήθελα από πλευράς μου να πω πόσο με ικανοποιεί το ότι οι συνάδελφοί μου αναγνώρισαν τον ιδιαίτερο ρόλο της Σουηδίας ε, ξέρετε ότι έχουμε πολλά δάση, μικρές ε, καλλιέργειες, τρεχούμενο νερό, ποτάμια, λίμνες. Ευχαριστώ τον Πάολο που παρευρέθη στην συνάντηση και συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό συζητήσει συζητήσεις μας. Για το θέμα του κλίματος, επίσης να αναφέρω άλλες δύο που έγιναν το φθινόπωρο στη Σουηδία. Ε, για το κλίμα και τα τρόφιμα, για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές τροφίμων και τι μπορούν να κάνουν για να μειώσουν την επιρροή που έχουν στο κλίμα. Στην άλλη διάσκεψη, ε, διαμόρφωση της, ε, του μέλλοντος της υπαίθρου, ε, είδαμε πώς η ανάπτυξη της υπαίθρου μπορεί να συμβάλλει τόσο ώστε η κοινωνία να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις του κλίματος. Παραδείγματος χάρη προαγωγή της περαιτέρω αηφόρου ανάπτυξης της βιοενέργειας. Ε, στο, στη Γεωργία ε, το φθινόπορο έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν και από την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των εξελίξεων στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής. Όπως είπα και το Σεπτέμβρη, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα και ξαναλέω ότι ήδη συνιστούσε προτεραιότητα για την Σουηδική Προεδρία. Αυξή... Αυξήθηκαν οι τιμές σχεδόν όλων των γεωργικών προϊόντων την περασμένη χρονιά και υπάρχουν ανησυχίες ε, κυρίως ως προς τους γαλακτοπαραγωγούς. Με τη σειρά του αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερη πίεση επί των Υπουργών για να κινηθούν σε πολιτικό επίπεδο και να αμβλύνουν τις δυσάρεσες επιπτώσεις της κρίσης στους γαλακτοπαραγωγούς. Συζητήθηκε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε ένα γεύμα που διοργανώσαμε συγκεκριμένα, ούτω ώστε να έχουν όλη την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διάλογο. Πολλά κράτη-μέλη ζήτησαν συγκεκριμένα μέτρα για σταθεροποίηση των τιμών και άμβλυνση ε, των δυσχεριών που προκύπτουν από την κρίση. Μετά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελικά τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, αποφασίσαμε να αναλάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε και μία ομάδα υψηλού επίπεδου που θα συνεχίσει να εργάζεται την Άνοιξη. Καλωσορίσουμε αυτόν τον νέο διάλογο. Είναι απαραίτητο ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό ο γαλακτοπαραγωγικό ε, τομέα. Είμαι πεπισμένο ότι οι εργασίε τη ομάδα υψηλού επίπεδου θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ στι γενικότερε συζητήσει σχετικά με το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Η γενική συζήτηση για την μεταρρύθμιση τη κοινωνική γεωργική πολιτική ε, φυσικά θα συνεχιστεί επί Ισπανική Προεδρία. Ε, το Δεκέμβρη 10 κάναμε και μία συζήτηση προς ανατολισμού σχετικά με την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Εκεί εστιάσαμε την προσοχή μα στο να εντοπίσουμε τι βασικότερε προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Γεωργία και τη Ευρωπαϊκή ανάπτυξη τη υπαίθρου και προσπαθήσαμε να δούμε με ποιο τρόπο τα προγράμματα ανάπτυξη υπαίθρου πρέπει να διαμορφωθούν ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τι προκλήσει. Ε, η συζήτηση είναι λογική απόρρια των συζητήσεων για τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο που οργανώσαμε το Σεπτέμβρη και όλα τα κράτη-μέλη Μίλησαν για αυτές τις τέσσερις βασικές προκλήσεις. Ε, προστασία του περιβάλλοντος, ε, ε, αηφόρος χρήση της ενέργειας και διατήρηση της βιοπικιλότητας και των υδάτινων πόρων. Αυτά είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου. Όταν ήρθα το Σεπτέμβρη συζητήσαμε για την ανάγκη που υπάρχει, την επιτακτική ανάγκη να γίνουν αλλαγές. Χρειάζεται να να κάνουμε αλλαγέ χωρίς όμως ε, να διωγγώσουμε το διοικητικό άχθο. Ε, και προετοιμα... Ε, παρουσιάσαμε συγγνώμη και τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 39 συγκεκριμένα μέτρα απλούστευση για την Ήπεθρο και είχαμε και μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση που μας επιτρέπει να δούμε πώς μπορούμε να απλουστεύσουμε την κοινή γεωρική πολιτική. Ε, το ίμιση των κρατών μελών ε, τελικά υπέβαλαν προτάσεις που θα ακολουθηθούν και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να είναι ευανάγνωστη και απλή και για τους γεωργούς, για τους χρήστε και για ολόκληρη την ε, κοινωνία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτική να νομιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την αγαστή συνεργασία που είχαμε επί Σουηδική προεδρία. Ε, με το Κοινοβούλιο γενικότερα και πιο συγκεκριμένα με την Επιτροπή σα για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και δοκιμές. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα της διαδικασίας συναπόφασης το οποίο επιλήθηνε το φθινόπωρο και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και ε, σας εύχομαι καλή τύχη για να καταλήξετε συμφωνία με το Συμβούλιο για τα ουσιαστικά ζητήματα της πρότασης. Τώρα η Ισπανική Προεδρία επιφορτίζεται με το καθήκον να συνεχίσει τις συζητήσεις για την προσαρμογή της πρότασης της νέες διατάξεις της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συμμετέχοντες, κυρίως το, την εισηγήτρια, την ε, κυρία Μπετ Γέγκλε, η νέα οδηγία είναι σημαντικό βήμα ώστε να επιτύχουμε καλύτερη προστασία των ζώων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουμε επίσης την ανταγωνιστικότητά μας στον επιστημονικό τομέα, τομέα της επιστημονικής έρευνας. Ε, σχετικά με την υγεία και το ευζήν των ζώων τώρα, η Προεδρείο μας ε, διοργάνωσε μια διεθνή διάσκεψη τον Οκτώβριο στην Ουψάλα Μεταξύ άλλων έγινε τελική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Προγράμματος Welfare and Quality, Ευζήν και Ποιότητα και οι Υπουργοί Γεωργίας έκαναν επικοδομητικότατη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα που σας είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Μεταξύ άλλων ε, η μελλοντική πολιτική για την καλή υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από εντατικέ ε, πολιτικέ διαπραγματεύσεις ε, καταλήξαμε σε συμφωνία το Δεκέμβρη στο Συμβούλιο σχετικά με τους κανόνες ε, για του εκτροφείς και για τις παραγωγικές μονάδες Επίσης ε, μιλήσαμε για τα δάση και την προστασία τους χωρίς όμως να δημιουργήσουμε περίτα διοικητικά άχθη και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας θα προκύψει μια ε, συμφωνία στα πλαίσια της διαδικασίας ε, συναπόφασης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και για την απασχόληση σε κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε και η φόρο παραγωγή ενέργειας σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, μπορούμε, ε, δεν θέλουμε να αντικατασταθεί το ξύλο με άλλα υλικά λιγότερο φιλικά ως προς το περιβάλλον. Ιδού λοιπόν φίλοι μου τα επιτεύγματα της Σουηδικής Προεδρίας ε, προσμένω στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε τώρα. Σας ευχαριστώ Πάολο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Έσκυλ για μια παρουσίαση ενδιαφέρουσα, με πάθος, με ισορροπημένα στοιχεία και ξέρετε ότι οι κλιματολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει πολύ τις εργασίες μας όλο αυτό το χρόνο και θα μας επηρεάζουν και στο μέλλον. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Γέγκελ θα μιλήσει πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κατά την ολοκλήρωση της θητείας σας βρίσκεστε εδώ και μας αναφέρετε ποιες, ήταν, ε, ποιες ήταν οι δικές σας προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας. Ε, επιστημιστική ασφάλεια, ε, κλίμα, η ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτά είναι τρία σημαντικά θέματα τα οποία πρόκειται να μας απασχολήσουν για πολύ καιρό ακόμα. Ε, άλλα ζητήματα όπως είναι η οδηγία για τις δοκιμές με τα ζώα, αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε επεξεργαστεί από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Ήταν μια έκθεση ε, σε σχέση με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, ε, προετοιμάζοντας τη διαδικασία αυτή. Και στο υπόβεθρο αυτό ασχοληθήκαμε με θέματα τα οποία δεν γνωρίζαμε πολύ καλά και μπορέσαμε να εργαστούμε πολύ καλά ε, και σε θέματα επί της ουσίας και να συνεργαστούμε με, την, ε, με τις περισσότερες από τις πολιτικές ομάδες και να πετύχουμε μια συνένεση, μια συμφωνία. Ήταν δύσκολο το θέμα αυτό, τα πειράματα με τα ζώα. Όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία των ζώων ε, παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες. Από την άλλη, τέλος, σημαντικά για μας ως πολίτες και ως βουλευτές. θεωρώ ότι και εσείς ως Σουηδός Υπουργός, γεωργίας ε, θα παραμείνετε ανοιχτοί προς τα ενδιαφέροντα του Κοινοβουλίου και θα ε, τίνετε δίκον για τις δικές μας προτάσεις και ιδέες τις οποίες θα μεταφέρετε ε, στη χώρα σας. Νομίζω ότι υπάρχει και από τις δύο πλευρές το ενδιαφέρον για μια συνέχιση της συνεργασίας αυτό θα είναι υπέρ τη ε, πολιτικής της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον υψηλό βαθμό διαφάνειας που πραγματικά ε, κυριάρχησε, πριτάνευσε κατά τη διάρκεια της θητείας. Σα ευχαριστούμε πολύ εσά προσωπικά και την εξαίρετη ομάδα σας. Ευχαριστώ Ελίζαμπεθ. Minister, ich auch ganz herzlich... Ε, ναι. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την εργασία σας. Ε, κυρία Γέκλε, ανέφερε τον υψηλό βαθμό διαφάνεια για τον οποίο φροντίσατε και διέκρινε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε τα θέματα. Και πραγματικά η δουλειά σα ήταν εύκολη σε μια εποχή όπου στη Γεωργία υπήρξε μια μεγάλη κρίση λόγω ακριβώς των τιμών, ιδιαίτερα στον γαλακτοκομικό τομέα. Και ε, τα προβλήματα λύθηκαν με επιτυχία και δείξατε ότι είστε ανοιχτοί στο διάλογο προς όλες τις πλευρές και ανοίξατε την πόρτα σε ανθρώπους που στο παρελθόν δεν είχε κανείς συμπεριλάβει στο διάλογο. Για το, λόγο αυτό θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε ε, θερμά. Επίσης, ε, επικεντρώστε την προσοχή σας στο πολύ σημαντικό θέμα της προστασίας ε, του περιβάλλοντος και της, σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό είναι ένα θέμα που θα σας απασχολήσει και στο μέλλον. Ε, δυστυχώς στη διάσκεψη της Κοπενχάγης ε, δεν έγιναν πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε το θέμα αυτό στην άκρη, αλλά ιδιαίτερα στο μέτρο της Γεωργίας θα πρέπει να ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής και πραγματικά να μένουμε με ανυπομονησία την αυριανή συζήτηση και πραγματικά μας δώσατε σημαντικά ερεθίσματα τα οποία θα συνεχίσουν να μας ασχολούν εδώ στους κόλπους αυτής της Επιτροπής. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας σηματοδοτεί μια νέα εποχή και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία μαζί με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον διάλογο και από κοινού να συμπεριλάβουμε πολλά θέματα. Καπούλα Σάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, θα ήθελα, προσωπώντα την ομάδα μου, αλλά και προσωπικά, να σε ευχαριστήσω για την Προεδρία σας. Ήταν ε, ήπια. Ε, χαρακτηρίστηκε από καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ασχοληθήκατε με μελλοντικά ζητήματα, κλιματικές αλλαγές, ε, με αξίες ε, που έχουν σχέση με το πολιτιστικό πρότυπό μας, το ευζήν των ζώων, το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας και κυρίω η φοβερή κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Μετά τον απολογισμό και το πέρας της Σουηδικής Προεδρίας, αυτό που μας ανησυχεί εμά τώρα στο Κοινοβούλιο είναι το άμεσο μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής της Ένωσης. Διάβασα τις ε, πρόσφατες δηλώσεις σας ε, για το πέρας του έτους ε, μετά από την διάσκεψη του Παρισίων όπου συμμετείχαν 22 κράτη-μέλη που υπερασπίζονται μια ισχυρή κοινή γεωρική πολιτική και άκουσα τις επικρίσεις που απευθύνατε σε αυτή τη σύσκεψη και εφόσον στο μέλλον η Σουηδία θα μας ε, βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια πιο ε, ίση και δίκαιη γεωρική πολιτική με τους πόρους που διαθέτουμε, θα θέλαμε στα πλαίσια του απολογισμού της Προεδρίας σας, που είναι θετικός κατά την άποψη όλων, θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε από τη Σουηδία στο άμεσο μέλλον, για αυτό το ζήτημα που τόσο μας ανησύχει, μεταρρύθμιση για την περίοδο δηλαδή μετά το 2013. Κυρία Χάουκεν, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω βαθύτατα την ε, Σουηδική Προεδρία. Βέβαια μια κάποια κριτική μπορεί κανείς να την κάνει προς την ε, Προεδρία αυτή. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το κλίμα στην Κοπενχάγη διαπιστώσαμε ότι οι Σουηδοί δεν ήταν ιδιαίτερα παρόντες ε, όταν συζητήθηκε το σημαντικό κατά τα άλλα θέμα της δασοκομείας. Ξέρετε ότι η Σουηδία έχει μια εθνική πολιτική και προασπιστήκατε τα εθνικά σας συμφέροντα. Το ίδιο έκαναν και άλλες χώρες ε, όπως η Αυστρία και η Φιλανδία. Αλλά ήσασταν η προοδρεύουσα χώρα και θα έπρεπε να τηρήσετε μια περισσότερο επικοδομητική στάση. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα των δασών θα έπρεπε ε, να συζητηθεί σε διεθνές επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια δυσκολία να παρουσιάσει στο θέμα των δασών μια ενιαία άποψη γιατί η Σουηδία ακολούθησε ένα αυστηρά προσωπικό δρόμο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν τα θέματα αυτά συζητήθηκαν στη Σουηδία και πώς θα μπορούσε η Σουηδία να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο και να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιαστεί με ενιαίο τρόπο και να μην ε, υπερασπιστεί με μειοπικό τρόπο τα εθνικά συμφέροντα που τη συναποτελούν. Υπάρχουν νέες δυνατότητες βραχυπρόθεσμης αλλά και μακροπρόθεσμης διαχείρισης πλέον των δασών. Δεν θέλω τώρα εγώ να αρχίσω μια τέτοια συζήτηση σε βάθος, αλλά έχω παρόλα αυτά την αίσθηση ότι στη Δανία ακολουθήσαμε μία γραμμή η οποία βασίζεται στην ιστορική μας εμπειρία ενώ η Φιλανδία και η Σουηδία ακολούθησαν μία αυστηρά οικονομική και εθνική ταυτόχρονα πολιτική. Και επίσης για τις υποανάπτυξη χώρες φυσικά δεν τους δώσαμε την προσοχή που θα έπρεπε. Λυπάμαι λοιπόν που δεν εφαρμόζονται οι τόσο προοδευτικές κατά τα άλλα θέσεις και στον τομέα των δασών. Καλώς. Κυρία Γκίνες. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σουηδική Προεδρία ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε σε μια ομάδα, ε, η αγοραστική δύναμη των ε, υπερκαταστημάτων, των σούπερ μάρκετς. Ξέρω ότι το θέμα αυτό απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Όταν ζητάμε από τους παραγωγούς να στρέφονται καλύτερα προς την αγορά, ε, και να προσαρμόζονται προς την αγορά ευκολότερα θα πρέπει και η αγορά να μην λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των παραγωγών. Διαρωτώ με λοιπόν πώς σχολιάζεται τη δύναμη που έχουν οι μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών σήμερα. Ευχαριστώ Μαγκίνε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ο επόμενος. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Έρλαντσον για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε τη Σουηδική περίοδο της Προεδρίας. Υπήρξαν πολύ περίπλοκα θέματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αυτής, όπως η παγκόσμια δημοσιονομική κρίση, η διάσκεψη της Κοπενχάγης, Υπάρχει ανάγκη να δούμε ακριβώς και με την κρίση η οποία χτύπησε τη Γεωργία κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιο είναι το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής μετά το 2013 οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν είναι επαρκείς, ήταν εύθετες χρονικά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τον Έσκιλ να ξαναπάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Παύλο. Αξιότιμοι βουλευτές, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Θα βάλω τα δυνατά μου για να συνοψίσω τις απαντήσεις που θέλω να δώσω στα σχόλια, της παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Ως προς τη συνθήκη της Λισαβόνας, πρώτα απ' όλα, θα έλεγα ότι η βασική θέση μας εν ώψη της Προεδρίας ήταν να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατό, ό,τι ήταν στο χέρι της Σουηδικής Προεδρίας, τόσο ώστε να ε, τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας αφοσιώσαμε και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί απίστευτα πολύ χρόνο και ενέργεια για να αρχίσει να ισχύει η συνθήκη Λισαβόνας διότι θεωρούσαμε ότι ήταν το καλύτερο για την Ευρώπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το εξής. Στις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου προωθούσαμε αυτή την στάση. Πριν τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης Λισαβόνας ε, προσπαθούσαμε να διεκπεραιώσουμε όλα τα ζητήματα ακόμη και αυτά που δεν αποτελούσαν αντικείμενο στην απόφαση προσπαθούσαμε να διεκπεραιώσουμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ως προς την προστασία των ζώων, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προασπίσουμε τα συμφέροντα των ζώων σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε γωνιά της Ένωσης να προστατεύονται τα ζώα και στο μέλλον θα αφιερώσω πολύ ενέργεια σε αυτό το θέμα για να έχουμε απτά αποτελέσματα για τις επιστημονικές δοκιμές με ζώα. Πέραν τούτου, μια άλλη ύψιστη προτεραιότητα της Προεδρίας μας ήταν να προετοιμάσουμε ε, το θέμα των κλιματικών αλλαγών εν ώψη της Κοπενχάγης. να από πλευράς γεωργίας ε, έχουμε πολλά να προσφέρουμε και σε σχέση με τα δάση μας. Στη Σουηδία επί μακρόν ακολουθούσαμε μια βιώσιμη δασοκομική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό. Δημιουργήσαμε οικονομική ευημερία σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ένωσης. Σήμερα Έχουμε ενεργειακή παραγωγή από τα δάση μας ε, που ανέρχεται στο 27% της ε, συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη Σουηδία. Και σήμερα βέβαια γνωρίζετε πόσο βιομηχανοποιημένη είναι η χώρα μας, άρα είναι υψηλό το ποσοστό. Είναι υψηλότερο και σε σχέση με άλλες χώρες, διότι εμείς έχουμε και το ψύχος και την υγρασία να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε περισσότερα δάση σήμερα ε, σε σχέση με οποιαδήποτε χρονική στιγμή του παρελθόντος. Μεγαλύτερες δασικές εκτάσεις λοιπόν σε σχέση με το παρελθόν και είναι ένα πρότυπο που θέλουμε να εξάγουμε προς την λυπή Ευρωπαϊκή Ένωση και προς ολόκληρο τον κόσμο, διότι οδηγεί σε οικονομική ευημερία, σε απασχόληση, ακόμη και σε αεροκατοικημένες ε, περιοχές και προασπίζει την ε, ε, βιοπικιλότητα και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και θα χρειαστεί να μας υποστηρίξετε και εσείς για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Αυτό το κάναμε ταυτόχρονα με την επίτευξη ενός άλλου στόχου. Συγκεκριμένα, να αποδώσουμε την δέωσα προσοχή στα προϊόντα υλοτομίας ε, που ε, εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της πολιτικής μας. Και ελπίζω επί Ισπανικής Προεδρίας το Συμβούλιο να συμφωνήσει με το Συμβούλιο ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι σχετικές συμφωνίες ε, διότι θα έχουμε καλύτερη απασχόληση, ευημερία, βιοπικελότητα και αντιμετωπίση της ε, παράνομης ε, υλοτομίας που παρατηρείται κυρίως σε άλλα μέρη του κόσμου. Ελπίζω στο μέλλον να τα καταφέρουμε. Eh, Τέλος. σε πολλούς ε, γεωργικούς τομείς υπάρχει μία αστάθεια. Επικροτώ δηλώσεις της Επιτροπής βάσει των οποίων ε, οφείλουμε να εξετάσουμε τους συσχετισμούς δυνάμεων για τον ανταγωνισμό, ε, μιλώντας για τα τρόφιμα. και επικροτώ την έκκλησή της προς τα κράτη-μέλη για να εξετάσουν ακριβώς ε, το, την ανταγωνιστική τους θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ε, είναι ευμετάβλητες ε, οι τιμές. Αυτό που παρατηρούμε σε πολλούς γεωργικούς ε, τομείς δεν είναι καλή η ανταγωνιστική μας θέση. Είτε μιλάμε για το στάδιο πριν το γεωργό, είτε για το επόμενο, της θέσεις εμπορία. Θα πρέπει να κατοχυρώσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα πριν και μετά το Γεωργό. Όμως εκείνος έχει την καταλητική δύναμη, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από ε, αυτούς, ε, διότι υπάρχουν πολλές σύνθετες πιέσεις στην αγορά μετά το στάδιο της καλλιέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση στην αγορά και με χαροποιεί το ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοινού τι μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Να αποφύγουμε την φθήνουσα κερδοφορία για τον παραγωγό και την αύξηση των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πάολο. Bene. Καλώ σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Ερλάνσον για την εξαιρετική εργασία της Σουηδικής Προεδρίας. Ε, θα διακόψουμε για ένα λεπτό να χαιρετήσω τον Υπουργό Έσκυλ. Μετά πάρτε τις κάρτες σας παρακαλώ γιατί θα ψηφίσουμε. Μετά τον χαιρετισμό του Υπουργού θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες.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

Έχουμε πολλές ψηφοφορίες να κάνουμε, έχουμε 200 τροπολογίες, έχουν κατατεθεί στην έκθεση του κυρίου, στη γνωμοδότηση μάλλον, του κυρίου Ταραμπέλα. Οι σκιώδεις εισηγητές έχουν συμφωνήσει σε μια σειρά συμβιβαστικών τροπολογιών και όλα αυτά θα μας βοηθήσουν στην ψηφοφορία να χαιρετήσω εδώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Τέστο από τη ΣΑΝΚΟ, την κυρία Νικολακοπούλου επίσης, πάντα από τη ΣΑΝΚΟ. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ταραμπέλα, από τον οποίο ζητώ να κάνει μια μικρή εισαγωγή πριν από το ξεκίνημα της ψηφοφορίας ευχαριστώντας τον για την προσπάθειά του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι φτάσαμε πράγματι σε μια καλή συνένεση. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες ε, τροπολογίες που δεν, στις δεν μπορούσε να επιτευχθεί συνένεση, αλλά θα υπάρξει μια δημοκρατική απόφαση. Ε, θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την ε, Επιτροπή. Ε, συμμετείχαν πάρα πολύ σε αυτό το ντοσιέ, το οποίο ενδιαφέρει Πολλέ πλευρές, πολλού ανθρώπους. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Λούλινγκ, τον κύριο Ράιμερ, τον κύριο Άσλινγκ, τον κύριο Νίκολσον, καθώς και τους βοηθούς τους. Επίση να τονίσω το ρόλο της ε, Γραμματείας για τη Γεωργία, ιδιαίτερα τον Όλιβερ Έμερ, ο οποίος ε, συμμετείχε ενεργά και επίσης του συνεργάτη μου Ζαμαρή Κουρτουά και Ζαν Ραμό που έκανε μια εργασία που πραγματικά ε, μας ε, απασχόλησε μέχρι την τελευταία στιγμή αλλά νομίζω ότι θα μας φέρει σε μια ε, ισορροπημένη λύση. Βεβαίως δεν θα μπορέσει να εικονοποιήσει όλες τις πλευρές αλλά νομίζω ότι πηγαίνει σωστή κατεύθυνση υπέρ των καταναλωτών κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική συνεργασία, το πνεύμα συνεργασίας που πριτάνευσε σε αυτή την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταραμπελά. Η κυρία Λούλινγκ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Ταραμπέλα. Ήταν ε, σχετικά εύκολο να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις, ούτως ώστε να έχουμε μία λογική έκθεση που θα οδηγεί σε μια εύκολα εφαρμόσιμη νομοθεσία χάρη στην οποία ε, μάλλον την οποία θα μπορέσουν όλοι εύκολα να εφαρμόσουν ε, ή με την οποία θα μπορούν να ζήσουν. Για την ε, συμβιβαστική λύση 2 δεν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ταραμπέλα. Ευχαριστώ την κυρία θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την 111. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία ψηφοφορίας θα πρέπει να κάνουμε ένα τεστ. <clears throat> Γι' αυτό σας παρακαλώ όλους να δοκιμάσετε την κάρτα σας να δούμε αν δουλεύει ή όχι παρακαλώ. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Καλώς κλείνει λοιπόν ο χρόνος ψηφοφορία. Η διαδικασία φαίνεται λειτουργεί και γι' αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είπαμε θα ξεκινήσουμε με την 111. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή η 111. 112. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται η 112. Περνάμε τώρα στην 16. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή η τροπολογία. 17. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. 113. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απερίφη. Η 114 τώρα. Α, όχι. Όχι, θα ψηφίσουμε την 114. Ξεκινάμε. Τέλος. Γίνεται δεκτή 114. 115. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. Απερίφθη. 116. Ψηφίζουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 18 τώρα. Ξεκινάμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Η 18 γίνεται δεκτή. 19. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 19 γίνεται δεκτή. Τροπολογία υπάριθμη 20. Ψηφίζουμε. Τέλος δεκτή 117 ψηφίζουμε τέλος απορρίπτεται 21 ψηφίζουμε ψηφίσατε όλοι Τέλος. Απορρίπτεται 21. Ερχόμαστε στην 118. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 118 απορρίπτεται. 119. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 22 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. 22 δεκτή. 23. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η 23 δεκτή. Η 120 ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Η 120 δεκτή. Η 121 τώρα. Ψηφίζουμε. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται η 121. Η 122. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται η 122. 123. Ψηφίζουμε. πέρα στις ψηφοφορίες Απορρίπτεται. 124. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 124 απερίφθη. 125. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 125 απορρίπτεται. 24. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Η 24 γίνεται δεκτή. Η 126 τώρα. Ξεκινάμε. Τέλος. 126 απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 25 δεκτή. Η 127 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 26. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται 26. 128. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή 128. 129. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Φτάνουμε τώρα στη συμβιβαστική πρόταση 1. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή η συμβιβαστική ένα. Προχωράμε τώρα και φτάνουμε στην 29. Ψηφίζουμε την 29. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Η 29 γίνεται δεκτή. 137. Ψηφίζουμε. Τέλος. Για 137 δεκτή. 138. Ψηφίζουμε. Τέλος δεκτή. 139. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η 30 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 140. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 140 απορρίφθηκε. Εκατόν σαράντα ένα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη. 143. Ψηφίζουμε. Τέλος. 143 δεκτή. 142 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 142 δεκτή. Η 31. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 31 δεκτή. Φτάσαμε τώρα στη δεύτερη συμβιβαστική. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή η δεύτερη συμβιβαστική. Περνάμε τώρα στην τρίτη συμβιβαστική. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή η τρίτη συμβιβαστική. Φτάνουμε τώρα στην τροπολογία 33. Ψηφίζουμε.

Δεκτή 154. Φτάνουμε τώρα στην 157. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή 157. Τώρα πάμε στην 162. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 162 απορρίπτεται. 163 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η 164 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος.

166. Ψηφίζουμε. Δεκτή. 167. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 168. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη. 169. Ψηφίζουμε. Τέλος. 169 δεκτή. 170 υπέρ. Τέλος. Απερίφθη. Α, για μια στιγμή. Δεκτή γίνεται η τροπολογία με μία ψήφο διαφορά. Τώρα 171 ψηφίζουμε. Τέλος. Η 171 δεκτή. 37, α όχι, έχει καταπέσει η 37. Πηγαίνουμε στην 172 Νικουλέσκου, ψηφίζουμε. Τέλος. Η 172 δεκτή. Τώρα φτάνουμε στην τέταρτη συμβιβαστική τροπολογία. Τέλος. Η συμβιβαστική πρόταση 4 γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στην 180. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 180 απορρίπτεται. 181. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη. 182. Ψηφίζουμε. Τέλος. για μια στιγμή έχουμε σημειώσει εδώ μία ψήφο επιπλέον. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 182. Έχουμε μία ψήφο επιπλέον από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρακαλώ να προσέξετε. Ψηφίζουμε εκ νέου λοιπόν την 182. Παρακαλώ να ψηφίσουν μόνο αυτοί που έχουν δικαίωμα. Ξεκινάμε. Τέλος. Η 182 απερίφθη. 184 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη και 184. Τώρα η 183. Ξεκινάμε. Τέλος. Δεκτή. Η 183 δεκτή. 39. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 39 γίνεται δεκτή. 185 τώρα ψηφίζουμε. Τέλος. Η 185 απορρίπτεται. Η 40 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 140 δεκτή. Η 40 μάλλον δεκτή. Τώρα περνάμε στην 186. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή 186. 187. Α, ξεκινάμε. Τέλος. Η 187 απορρίπτεται. Η 191 υπέρ. Κλείνουμε. Η 191 δεκτή. 193 τώρα ψηφίζουμε. Τέλος. Η 193 δεκτή. Τώρα περνάμε στην συμβιβαστική τροπολογία υπαρίθμων 5. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή η πέμπτη συμβιβαστική. Φτάνουμε τώρα στην τροπολογία 43. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 43 απορρίπτεται. 202. Ψηφίζουμε για τη 202. Τέλος. Δεκτή. 203. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 44. Υπε... Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 204. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 204 απερίφθη. Πηγαίνουμε τώρα στην 210. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 210 δεκτή. Η 211. Ξεκινάμε. Τέλος. 211 δεκτή. 45. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 45 απερίφθη. 212. Ψηφίζουμε. Τέλος. 212 απορρίπτεται. 214 τώρα ψηφίζουμε. Τέλος. Η 214 απορρίπτεται. 216 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 215 ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 46. Ψηφίζουμε. Κλείνουμε. Δεκτή. 213. Ψηφίζουμε. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Η 213 απορρίπτεται. 219 Lion. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή 219. Πηγαίνουμε τώρα στη 220. Ψηφίζουμε τη 220. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη 220. 221. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη 221. 48. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 48 απερίφθη. Τροπολογία 49. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 49 δεκτή. 50. Α, η 50 έχει αποσύρθει. Τώρα περνάμε στη 222. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 222 απερίφθη. 223. Ψηφίζουμε. Τέλος. Τώρα πάμε στην έκτη συμβιβαστική τροπολογία. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η έκτη συμβιβαστική. Τώρα περνάμε στην έβδομη συμβιβαστική. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. Τώρα ψηφίζουμε την 227. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή η 227. 229 Μαγκίνες ψηφίζουμε. Τέλος. Η 229 γίνεται δεκτή. 230. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 230 δεκτή. Η 51 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 51 απορρίπτεται.

Απερίφθη 2.34. Ψηφίζουμε τώρα την 53. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Δύο τριάντα πέντε. Ψηφίζουμε. Η 2.35 λοιπόν απορρίπτεται. 54. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και η 54. 236. Ξεκινάμε. Τέλος. Δεκτή. 2.37. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται η 2.37. 2.38. Α, είναι ταυτόσημη. Πηγαίνουμε λοιπόν τότε στην 240. Ψηφίζουμε. Τέλος.

και γι' αυτό πηγαίνουμε στην 56. Ψηφίζουμε για την 56 παρακαλώ. Τέλος. Δεκτή. 246 τώρα. Ψηφίζουμε. 246. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 247 ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 248 ανοιχτή διαδικασία. Κλείνει η διαδικασία. Απορρίπτεται. 57. Ψηφίζουμε. Θέλετε να την αποσύρουμε. Λοιπόν, η 57 απεσύρθη. Ψηφίζουμε τώρα την 249. Έχει αποσυρθεί και η 249. Κύριο Ταραμπελά έχει ζητήσει το λόγο. Στην αρχή είχα ενδιασμούς ε, για αυτό το θετικό σημάδι που φαίνεται θελκτικό, αλλά ξέρετε φοβούμε ότι Υπάρχει και ένας κίνδυνος, ξέρετε ότι είμαι τελείως αντίθετος, δηλαδή τι να μιλάμε για χαμηλές θερμίδες ενώ εγώ υπερασπίζομαι προϊόντα που μπορεί να μην είναι και τόσο υποφελή για την υγεία, αλλά εν περιπτώσει μπορούμε να τα καταναλώνουμε σε μικρές ποσότητες. Γι' αυτό υπέβαλε εγώ αυτή την τροπολογία, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, θα την αποσύρω. Ευχαριστώ. Τώρα είμαστε στο 249. Ψηφίζουμε για το 249 παρακαλώ. Τέλος. Δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην 261. Ψηφίζουμε τη 261. Επαναλαμβάνω, κάνουμε ένα άλμα και φτάνουμε στη 261. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Uh, uh, Έχω μια σύγχυση εδώ. Εγώ ψήφισα με τον ένα τρόπο στη μία ψηφοφορία και με διαφορετικό στην άλλη και τώρα έχουμε επανέλθει πίσω. Μήπως υπάρχει ε, πρόβλημα με τις δύο τελευταίες ψηφοφορίες παρακαλώ. Την 261 και την 61. Κοιτάξτε, ψηφίσαμε τη 261 κανονικά, γιατί έχοντας εγκρίνει την προηγούμενη τροπολογία, αυτόματα περνάμε στην 261. Εγκρίναμε λοιπόν την 261 και τώρα συνεχίζουμε με την 264. Εντάξει. Λυπάμαι άλλαξα την ψήφο μου. Γιατί είπατε ότι θα ψηφίσουμε την 61. Και μετά είπατε 261. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια σύγχυση και με επηρέασε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ η 261 να ψηφιστεί εκ νέου. Ε, ε. Non cambia comunque. Όχι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και ο Βαν Όρντεν χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούσαμε τι λέει. Κοιτάξτε, αν δει κανεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 261 που είναι ακόμα στην μικρή οθόνη, δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη αλλαγή. Και δεν μπορούμε εμείς να ξανακάνουμε εκ νέου την ψηφοφορία. Είναι θέμα κανονισμού. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε εκ νέου. Θα συνεχίσουμε και πηγαίνουμε στη 264. Παρακαλώ θέλω την προσοχή σας. Τελείωσε η 261, δεν ξαναψηφίζεται. Περνάμε τώρα στην 264. Κράιμερς, ψηφίζουμε. Για την 264 ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφη 264. Τώρα πηγαίνουμε στη 265. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 265 δεκτή. 266 τώρα. Ψηφίζουμε. 266. Τέλος. Απερίφθη. Α, για μια στιγμή. 2.67 τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 269. Φτάνουμε τώρα στο 269 Lion. Ψηφίζουμε την 269. Τέλος. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 64. 64. Ψηφίζουμε Τέλος. Δεκτή. 65. Ψηφίζουμε την 65. Τέλος. Δεκτή. 66. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 66. Τέλος. Δεκτή. 67. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 67 δεκτή. 68. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 68 δεκτή.

Ψηφίζουμε τώρα την 70, τροπολογία 70. Τέλος. Η 70 δεκτή. Η 71. Ξεκινάμε. Τέλος. Δεκτή η 71. 72. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 2.72 τώρα. 2.72. Τέλος. Δεκτή. 73. Ψηφίζουμε. Τέλος.

Τέλος. Η 273 περίφη. 274. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 275. Τέλος. Δεκτή 275.

277. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 277 δεκτή. 278. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 279. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 2.80. 2.80. Τέλος. Απορρίπτεται. 2.81. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 2.81 δεκτή. 2.82. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 282 δεκτή. 283 ψηφίζουμε. Τέλος. 283 απορρίπτεται. 284 ψηφίζουμε. Τέλος. 284 δεκτή. 285 ψηφίζουμε. Τέλος. 285 απερίφθη. Παρακαλώ πρέπει να ψηφίζουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία. 286. Ψηφίζουμε. Τέλος. 286 δεκτή. 288. Ψηφίζουμε. Τέλος. 288 δεκτή. Έχουμε επίσης και την προφορική τροπολογία Gladfelder. Συμφωνείτε να την ψηφίσουμε. Του δίδω το λόγο. Η ε, η χρήση συγγνώμη, του όρου μέλη στον προσδιορισμό του προϊόντα ή ε, οποιοδήποτε γραφικό ή μη γραφικό στοιχείο, ε, γραφίστικο ή μη γραφίστικο στοιχείο, το οποίο είναι μία ένδειξη ότι το προϊόν περιλαμβάνει μέλι ή τα 50% του προϊόντος προέρχονται από μέλι. Λοιπόν, ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία Gladfelder. Ψηφίζουμε. Segnale. Chiuso Δεκτή η προφορική Gladfelder. Περνάμε τώρα στη 287. Γέγκλ. 287. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 77. Ψηφίζουμε την 77. Τέλο. Δεκτή. 78. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 79. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 80. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 81 ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 289 αντελάγκε. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 289 δεκτή. 82. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 2.90. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 2.91. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 2.91 δεκτή, 2.92 ψηφίζουμε. Τέλος. 292 δεκτή. 293 ψηφίζουμε. Τέλος. Η 293 δεκτή. Και στο τέλος 83. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 83 δεκτή. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει αρκετά. Τελειώνουμε όπου να με. Περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Η 85. 85. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή η 85. Η 87 του Λαβία. Ψηφίζουμε. Τέλος. 88. 88 κατά ψηφοφορία εδώ. Το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Τέλος το πρώτο τμήμα. Δεκτό. 88 δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτό και το δεύτερο τμήμα. 89. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτό. Τροπολογία υπαρίθμ 2. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη. 4. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η 90. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η 5. Ψηφίζουμε. Τέλος. Η 5. Δεκτή. Η 91. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας για την 91 απερίφθη. Τροπολογία υπαρίθμ 6. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Τελευταία σελίς. Τροπολογία 7. Ψηφίζουμε. Τέλος δεκτή. 92. Α, όχι. 92 έχει καταπέσει πλέον. Η 8 πλέον. Ψηφίζουμε την 8. Τέλος. Δεκτή. Η 94. Ψηφίζουμε. Τέλος. Πάλι έχουμε μία ψήφο επιπλέον από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει κάτι λέει ο Πρόεδρος, αλλά σας παρακαλώ πολύ να ψηφίζουμε αυτοί που πρέπει. Περνάμε τώρα στην 96. Ψηφίζουμε την 96. Τέλος. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για το 96. Πάντα υπάρχει ένας επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για το 96. Τέλος της ψηφοφορίας για την 96. Δεκτή η 96. Περνάμε στην 10 τώρα. Ψηφίζουμε την 10. Τέλος. Πάντα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ένας επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. 10. Siamo al 10. Dobbiamo ripetere. Ripetere. poi andiamo. Grazie Albert. Ευχαριστώ Άλμπερτ. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία υπαρήθμ 10. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η 102 τώρα. 102 Ντελάνγκε. Ψηφίζουμε. Τέλος. Ο Ντες έχει δει το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ε, κάτι εδώ δεν μπορεί να ισχύει. Δύο τακτικά μέλη δεν είναι παρόντα και ψηφίζει μόνο η Άστριτ Λούλινγκ ως αναπληρωματικό μέλος. Δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι ψήφοι.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 Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την 102, 102, Ντελάγκε. Κοιτάξτε, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να σηκώσουν το χέρι τους. Παρακαλώ, δεν πρέπει να είναι άνω των 17. Ποιοι ψηφίζουν για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σηκώστε το χέρι σας. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sind zwei hinten in der Okay, Reihe. 18. 18. Ja. Okay. Per favore. Λοιπόν, μόνο αυτοί που σήκωσαν το χέρι ψηφίζουν. Κανείς άλλος παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε για μια ακόμη φορά την 1-0-2. Τέλος. Απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα την 12. 12. Τέλος της ψηφοφορίας για την 12. Δεκτή. Η 108 τώρα. 108 Νίκολσον. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απερίφθη. 13. Ψηφίζουμε για την 13. Τέλος. Απερίφθη. 14. Ψηφίζουμε για την 14. Τέλος. Δεκτή 14. 15. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. 109. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Και τώρα η τελική ψήφος. Τελική ψήφος παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Και εδώ τελειώσαμε. Νομίζω ότι καλά πήγα λέει ο πρόεδρος εκτός από μια στιγμή όπου κάπου τα χάσα. Prego di prendere posto. Παρακαλώ, καθίστε. Δεν έχουμε τελειώσει. Otherwise we are long time. Stefan. Se vuoi metto la mano, così urlo quando... Madame Paulson.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 Valutazione del bilancio del programma d'azione comunitario. Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης. Dura e benessere degli animali. Για την ευημερία των ζώων παρακαλώ πρέπει να καθίσετε. Έχουμε αρκετή δουλειά. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της ευημερίας των ζώων και ευχαριστώ τον κύριο, την κυρία Πόλσον η οποία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η σωστή φροντίδα των ζώων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ε, γεωργίας, της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και της σύμπανσης. Το 2006 η κυρία Γέγκλε συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση που αποτέλεσε στη συνέχεια έρισμα για τις μελλοντικές εργασίες ε, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου τα τελευταία έτη. Τώρα Οι απαιτήσει του Κοινοβουλίου και της κυρίας Γέγκλε δεν έχουν πληρωθεί. Πόρο απέχουμε. Καλύπτουμε ζητήματα όπως τα πειράματα με ζώα που, στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα και άλλα θέματα σχετικά με τη φροντίδα των ζώων που εμπλέκονται και στις διαπραγματεύσεις ε, του ΠΟΕ σε ένα ορισμένο βαθμό. Έχουμε σημειώσει βήματα προόδου, αλλά υπολείπεται σκληρό έργο βάσει του προγράμματος που συντάξαμε το 2006. Και στο ψήφισμα το Κοινοβούλιο επέμεινε ότι έπρεπε να χρησιμοποιούμε τις βέλτιστες μεθόδους και επιστημονικές γνώσεις για τη σύνταξη ενός πενταετούς σχεδίου. Αυτό το πενταετές σχέδιο δρομολογείται φέτος. Το σημαντικότερο είναι το τι έπεται, το νέο σχέδιο. Συμμετείχα στα θέματα της επιστημιστικής ασφάλειας, ασφάλειας των τροφίμων και της ευημερίας των ζώων σε συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία 7 χρόνια και έχω κουραστεί πλέον. Κάθε 5 χρόνια οι οργανώσεις των φίλων βγάζουν αυτά τα πέσια φιλμ για τα ζώα και παρουσιάζουν αυτή την ιδεχθή εικόνα στους καταναλωτές. Φυσικά όλοι νιώθουμε αποτροπιασμό και νομίζω ότι τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να συζητάμε τα θέματα ηθικής, δεοντολογίας ε, και το δικαίωμα των ζώων για μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα. Τι γίνεται στην πράξη. Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί τώρα η οικονομία μας. Γίνεται τώρα να συγκροτήσουμε ένα ορθό σύστημα προστασίας των ζώων που να μπορούν τώρα να εφαρμόσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη η γεωργία και εκτροφής. εκτροφείς. Μπορώ να σας δώσω άπειρα παραδείγματα σχετικά με το ανέφικτο του εγχειρήματος. Απαγορεύει λόγου χάρη η Σουηδία τα μη διευθετημένα κλουβιά για τις ε, ο παραγωγές, ε, ο παραγωγούς όρνηθες και τελικά τι γίνεται, μετατοπίζεται η εκτροφή στη Φινλανδία. Και κανείς δεν αγοράζει αυγά από εκτρεφόμενες ε, όρνηθες. Και η βιομηχανία τι κάνει, στρέφεται προς τα φθηνότερα αυγά. Προτείνω λοιπόν αφενός να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό επίπεδο για όλα τα κράτη-μέλη, για όλες τις περιφέρειες, για όλους τους εκτροφείς. Όλοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με κοινά πρότυπα. Εάν δεν έχει συμμορφωθεί κανείς, δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα θέση εμπορία ζωικών προϊόντων. Μόνο έτσι μπορούμε να αναχαιτήσουμε τις εισαγωγές από χώρες που δεν επιβάλλουν τις ίδιες απαιτήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντική πρόκληση αυτή των, ε, του ισότιμου ανταγωνισμού των ομοιόμορφων προτύπων για όλους τους παραγωγείς. Ε, αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Κοινή νομοθεσία, λοιπόν, μέσα στην έκθεση επεξηγώ όλα όσα σχετίζονται με την σχετική νομοθεσία που έχει εκπονηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει ε, λειτουργήσει με εξαιρετικό τρόπο το σύστημα. Το μόνο που δεν λειτουργεί είναι η συμμόρφωση με τα νομοθετήματα. Και αυτό θα έχει την καταλητική σημασία. Οφείλουμε να έχουμε ένα σύστημα, αλλά και να ελέγχουμε την συμμόρφωση προς την νομοθεσία. Λυπούμε που το λέω, αλλά για να λειτουργήσει σωστά ένας νόμος πρέπει να υπάρχει και σύστημα ποινών που το συνοδεύει. Και αυτό είναι το επόμενο σημείο κρίσιμης σημασίας. Κατόπιν, η σχέση ανάμεσα στην υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία. Άλλο σημαντικό ζήτημα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά επικίνδυνες νόσους και αναπτύσσουμε πολυανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά και τα ζώα και οι άνθρωποι. Αυτό είναι πραγματικά υπέρμετρα ανησυχητικό. Με την προστασία των ζώων αυξάνεται η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Αυτό έχει ε, κέρια σημασία και για την υγεία των ζώων και για τη δημόσια υγεία. Ελπίζω να διαβάσατε όλη την πρότασή μου και ελπίζω ότι με αυτές τις δύο προτάσεις που έκανα επί της αρχής θα συμφωνήσετε και αυτή τη σχέση με την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά και τη σχέση με τη δημόσια υγεία. Κατά τα λοιπά, μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά ελπίζω, έλεγα, ότι θα συμφωνήσετε με τις βασικές αρχές. Και κυρίως να συμφωνήσουμε όλοι για την αρχή ότι πρέπει να υπάρχουν παντού ομοιόμορφες απαιτήσει, οι ίδια δικαιώματα, όλοι πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσης όρης ε, από οικονομικής ε, πλευράς. Ε και αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε πρόκειται για εκτροφής, είτε πρόκειται για παραγωγούς ζώων συντροφιάς. Στην πράξη, τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να υλοποιήσουμε ε, ένα ε, λογικό νομικό και εκτιμένο, εύκολα εφαρμόσιμο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Παουλσένε, πριν αρχίσουμε την συζήτηση, ας ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Γκαρινέλη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσεν και την Επιτροπή σας για τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε σχετικά με το θέμα της προστασίας των ζώων. Είναι προτεραιότητα το θέμα του ευζήν των ζώων για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά άμεσα επίσης και την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να δούμε τι έχουμε πετύχει σε σχέση με το πρόγραμμα των τελευταίων 10 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό μια πολιτική αξιολόγησης της προστασίας των ζώων τα τελευταία 20 χρόνια. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από διάφορους εμπλεκομένους ευρωπαϊκούς φορείς και θα ολοκληρωθεί προβλέπεται το Δεκέμβριο του ενεστώτος έτους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής μαζί με την έκθεσή σας θα είναι ένα βασικό βήμα θα έλεγα για τον καθορισμό των νέων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλώς ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Πρέγω θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πάουλσεν την εξαίρετη εργασία τη σε αυτό το τομέα και για την προσέγγιση που παρουσιάζει εδώ. Κυρίω στο πρώτο τμήμα τη έκθεση της. Βεβαίω βασιζόμαστε στην εργασία που έχει γίνει ήδη στην προηγούμενη θητεία και νομίζω ότι έχουμε ήδη κάνει κάποια βήματα προς τα μπρος όσον αφορά τη βελτίωση της ευημερίας των ζώων. Αλλά βεβαίως απομένουν πολλά πράγματα να γίνουν. Και όπως και η κυρία Πόλσεν αναφέρει, δυστυχώς πολλές από αυτές τις ιδέες ε, παραμένουν ακόμα στα χαρτιά. Και είναι σαφές ότι η κατάσταση επιδέχεται βελτιώσεων. Όσον αφορά το πρόβλημα αυτό σαν μια πρόκληση προς την ανθρωπότητα θα έλεγα, γιατί δεν είναι το ζητούμενο να βάλουμε το κέρδος ε, μπροστά από την ευημερία των ζώων. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ως ανθρώπινα όντα δεν θα πρέπει να είμαστε βάναυση προς τα ζώα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου, όχι μόνο στις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, αλλά και τις σχέσεις με τα ζώα, γιατί είναι ένα μέτρο της ανθρωπότητας. Έχοντας ακούσει την εισαγωγή της κυρίας Πόλσεν, θα ήθελα απλώς να πω ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι θα πρέπει να τηρήσουμε υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ευημερία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε την εικόνα των εισαγωγών και εξαγωγών. Θα πρέπει να δούμε πώς, ε, ποια είναι η απόδοση των παραγωγών μας εντός της κοινότητας και εκτός αυτής. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε παράγει κάτι, παράγει ζωικά προϊόντα στην επικράτεια της κοινότητας, είτε για την εγχώρια κατανάλωση, είτε για την εξαγωγή, θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές μπάση περιπτώσει. Με τον ίδιο τρόπο. Και για τις αγωγές και για τις εξαγωγές. Δεν θα πρέπει να προεξάρχουν οι καθαρά αυστηρά εμπορικοί υπολογισμοί. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εμπεδώσουμε αυτές τις αρχές. Ελπίζω ότι η κυρία Πόλσον ως συγγήτρια θα έχει κατά νου και κάτι άλλο. Δηλαδή ότι έχουν γίνει βεβαίως πολλές συνεδριάσεις και υπάρχει το Intergroup για την προστασία των ζώων και έχουν διατυπωθεί κάποιοι κανόνες μεν, αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα όσον αφορά την πλευρά της ε, εφαρμογής. Γιατί ε, έχουν γίνει πολλές ε, δηλώσεις έχουν διατυπωθεί κάποια κριτήρια, αλλά δεν εφαρμόζονται πάντοτε. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική εποπτεία στο επίπεδο των χωρών μελών, πιστεύω. Νομίζω ότι αληθεύει να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πτυχή της εφαρμογής στην πλειονότητα των χωρών μελών. Και από αυτό εξαρτάται ε, ε, και η ποιότητα της ευημερίας των ε, ζώων η, ποιότητα των ελέγχων ε, εξαρτάται από την ε, αξιοπιστία των ελεγκτικών, των εποπτικών οργάνων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για μια κατάλληλη ε, αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων. Γιατί πάντοτε υπάρχουν κάποια χάσματα εδώ και να. Η έκθεση της κυρίας ε, Πόλσον ε, δεν θα πρέπει να μπει απλώς ε, στο χαρτοφυλακά μας, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη σωστής εφαρμογής. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βετσαχόφσκι. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 9 Φεβρουαρίου 12 η ώρα. 9 Φεβρουαρίου 12 η ώρα είναι η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών. Ο επόμενος η επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Γκαρθία Πέρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσεν για την εργασία τη σε αυτή την έκθεση. Αλλά θα ήθελα να κάνω καταρχήν μια παρατήρηση γενική φύσεω και στη συνέχεια να επισέλθω σε ειδικότερα θέματα σε σχέση με ορισμένα σημεία τα οποία εισάγει η έκθεση και που ελπίζω ε, ότι συν χρόνο ή μάλλον μέχρι την προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια κοινή θέση όσον αφορά ορισμένα βασικά ζητήματα. Ο κανονισμός για την ευημερία των ζώων θα πρέπει να εξελιχθεί πάνω σε μια επιστημονική βάση. Έχουμε μια νομοθεσία και ανακύπτουν το προβλήματα. Το πρώτο είναι να τα αναγνωρίσουμε και να τα απειλήσουμε πριν προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Ε, εάν δεν εφαρμόζεται θα πρέπει να ενεργήσουμε αυστηρότερου ελέγχου. Αλλιώ θα αναπραχθούν τα ίδια προβλήματα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανταγωνιστικότητα των πραγών. Έχουμε κάποια, κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές που συνεπάγονται ένα πλέον κόστος για τους παραγωγούς. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε τον τρόπο που θα τους αποζημιώσουμε. Ε, εάν ο καταναλωτής δεν πληρώνει αυτό το επιπρόσθετο κόστος, θα πρέπει να εξεύρουμε τις αντισταθμίσεις για τους ε, παραγωγούς και θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα όσον αφορά τις εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τώρα, όσον αφορά το σημείο 5, θεωρώ ότι η διατύπωση «λυπάται» δεν είναι δεδειγμένη. Ε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει προτάσεις, γιατί μέχρι στιγμής δεν διαθέτει μια νέα επιστημονική βάση, στην οποία ευαισθούν οι προτάσεις, οι οποίες να πηγαίνουν παραπέρα από αυτό που υπάρχει ήδη. Όσον αφορά το σημείο 7, νομίζω ότι δεν ενδείκνυται να ζητήσουμε από την Επιτροπή να ε, πληρεί τους ε, νόμους Ε, με αναφορά μόνο στις ε, οτόκες όρνηθες. Όταν γίνεται αναφορά στο σημείο 12 για τα ζώα, τι σημαίνει αυτό. Ότι η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ασχοληθεί με την ευημερία των ζώων, όσον αφορά τα ζώα συντροφιά κλπ. Ποιο ε, θα ελέγξει την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σκυλιά ή τα γατιά, τα κατοικίδια γέννη. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Νομίζω ότι στο 12 θα πρέπει να συμπελάβουμε τη διατύπωση εκούσια. Ε, Όσον αφορά το 16 έως το 18 ανακύπτει το θέμα, το θέμα ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ευημερία των Ζώων. Ποιος θα το πληρώσει όμως. Ήδη έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να δώσουμε στις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν ε, τις ε, δυνατότητες να πληρούν, να του στόχου για του οποίου έχουν συσταθεί και όχι να προβαίνουμε στη δημιουργία νέων Ινστιτούτων, νέων εργαλείων που συνεπάγονται αύξηση του κόστου και ε, εν γέννη θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ήδη φυστάμενους μηχανισμούς. Όσον αφορά το 24 έως το 28 ε, τις νομοθετήσεις ε, για την ευημερία των ζώων, αν φέρεστε στα αντιβιωτικά. είναι σαφές ότι οι κτηνίατροι δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Εδώ έχει ένα λόγο και η ιατρική. Οι ιατροί μάλλον. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξελίξει την δική της εργασία. Δεν είναι δική μας ευθύνη εδώ. Θεωρώ ότι μέχρι την, ε, μέχρι την ψήφιση της έκθεσης ε, θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία ε, επί πολλών σημαντικών σημείων. Ευχαριστούμε πολύ. Η εξάτιμη κυρία Ελίζαμπεθ Γέγκλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Οι πρώτες μου ευχαριστήσει απευθύνονται στην κυρία Πάουλσιν για την έκθεσή της και επίσης για την ειλικρίνεια με την οποία θέτει το θέμα εδώ. Το συζητούμε για δεύτερη φορά το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την προλαλήσασα ε, και θα ήθελα να το τονίσω ρητά εδώ. Έχω την άποψη ότι ε, πρόκειται να υποβάλουμε εν το συνόλο μια καλή πρόταση. Από τη δική μου πλευρά η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας θα πρέπει να θέσει το επίκεντρο στην αξιολόγηση αυτού που έχει συμβεί από το που έχει γίνει μάλλον από το 2006. Και εδώ αποσιάζουν βασικές πληροφορίες. Έχουμε θέσει υποβάλει κάποια αιτήματα, ε, ορισμένα έχουν εφαρμοστεί, αλλά όχι ορισμένα πράγματα έχουν εφαρμοστεί στις χώρες μέλη, άλλες στις χώρες υπολείπονται στην εφαρμογή. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να επικεντρώσουμε στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης στο πώς ε, μπορεί κανείς να αξιολογήσει την εξέλιξη από το 2006 έως σήμερα και ποια είναι τα αιτήματα που θέτουμε επί τη βάση αυτής της αξιολόγησης. Ένα δεύτερο σημείο αφορά στην ε, λεγόμενη προστασία των ζώων. Εάν επατούμε κάτι τέτοιο, και θα ήθελα να θυμίσω τα όσα είπε ο κ. στην αρχή, η προστασία των ζώων βεβαίως θα πρέπει να ισχύει. Έχουμε τα πειράματα με τα ζώα και έχουμε και τα ζώα τα οποία χρησιμοποιούνται στην ε, γεωργία. Αλλά όταν μιλάμε Γιάννους για μας ως ανθρώπους ή για την κοινωνία συνολικά, στην έκθεση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί το αίτημα τα κατοικίδια ζώα να βρουν επίσης τη θέση τους εδώ, να αναφερθούν. Έχουν σημειωθεί πρόοδοι και ρωτώ τον κύριο Γκαρβινέλη που νομίζω είναι διατεθειμένος να μου απαντήσει. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, πρόοδοι ε, στις διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ. Ο κύριος με τον κύριο Γκαρδινέλη υπάρχει μια συνεργασία για το 2006 και κάποτε μου είπετε ε, όταν μου είπατε τι γίνεται όταν η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει ε, κάποια μέτρα για την προστασία των ζώων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολύ συχνά λέμε ότι εμείς θα πρέπει να λειτουργούμε σαν παράδειγμα για τους άλλους. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Έχει πράγματι τέτοιου είδους θετικές συνέπειες αυτή η δική μας παραδειγματική στάση. Τώρα, ε, τα ζώα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ε, νομίζω ότι εδώ χρειαζόμαστε μια στέρεη επιστημονική βάση. Μόνο σε αυτή τη βάση μπορούν να διενεργηθούν οι έλεγχοι. Νομίζω ότι στους ε, κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί μέχρι στιγμής και αναφέρεστε κυρία Πάουλσεν στους χείρους την έκθεσή σας, ε, εδώ υπάρχουν οι κανονισμοί της ΕΦΣΑ. Ε, δεν ξέρω, είναι επαρκής ή όχι. Θα, ή θα πρέπει να διαδεχθούν κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι αυτό, θα πρέπει να θέσουμε αυτό το θέμα, όπως και το θέμα της εφαρμογής μέχρι στιγμή στο επίπεδο των χωρών μελών. Εάν το πράξουμε τότε, νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και την Επιτροπή στον έργο της στο έργο της. Και είμαι σίγουρη ότι και η Επιτροπή καθώς και χώρες μέλη θα μας συνοδεύσουν με θετικό τρόπο από τη μία πλευρά ε, ε, θέσουμε το ζήτημα της προστασίας των ζώων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων από την άλλη και κατά τρίτο λόγο την προστασία όλων των ζώων συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιδίων. Ε, θα ήθελα να πω ότι μετά από αυτή την αρχική συζήτηση θα πρέπει να περάσουμε στο ε, θέμα της βελτίωσης λειτουργίας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με συγητή το Ζωζέ Μποβέ. Γι' αυτό παρακαλώ να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος και θα ξεκινήσω καταρχήν χαιρετίζοντας την έκθεση της ε, κυρίας Πόλσεν. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η υπόδειξή της για να υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές και κοινοί κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο, νομίζω ότι την ορθή προσέγγιση. Είχαμε, τέτοιες, ε, είχαμε εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών στη δική μου χώρα και όλοι έλπιζαν ότι θα υπάρξει μια βελτίωση της ευημερία των χείρων. Τελικά εξήχθη η παραγωγή σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν μια κοινή προσέγγιση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Τα άλλα δύο στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις κυρώσεις σε όλη την Ευρώπη ε, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι μία από τις μεγάλες αντιναμίες που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τις προδιαγραφές της ευημερίας των ζώων. Όσον αφορά τη μεταφορά, υπάρχουν νέοι κανόνες για τη μεταφορά εδώ και ένα χρόνο. Αλλά το θέμα δεν είναι οι νέοι κανόνες, αλλά η συμμόρφωση με τους κανόνες και η σωστή εφαρμογή τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά ε, το εμπόριο άλλων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η κοινή εφαρμογή θα πρέπει να ισχύει και για τις τρίτες χώρες και νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι θεμελιώδες. Εάν θέλουμε να προσπαθήσουμε ε, πράγματι να βελτιώσουμε την ευημερία των ζώων. Ε, χαιρετίζω επίση την ευκαιρότητα να έχουμε μια σωστή συζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι, κοινές, ε, ότι η κοινή εφαρμογή και οι σωστές και οι κυρώσεις είναι ο ορθός δρόμος. Ευχαριστώ. Με τη συνάδελφό μας Πινόζα, αύριο θα συζητήσουμε και το θέμα της αμοιβαιότητας των κανόνων. Ε, κυρία Μακίνες, ε, παρακαλώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια πριν περάσω στην έκθεσή σας. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι που έχουν κατοικίδια και εκτροφείς που φροντίζουν τα ζώα τους, έτσι. Βλέπουμε αυτές τις αποτρόπες εικόνες, αλλά δεν δίνουμε σημασία στα δυτικά παραδείγματα. Πρέπει να ε, υπερασπιστούμε και αυτούς τους εκτροφείς και τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων που ε, προστατεύουν τα ζώα. Μιλούμε συνέχεια για τη μία μειοψηφία. Δεύτερον, ξέρετε ότι ορισμένοι έχουν προβλήματα πνευματικής υγείας. Αυτοί βασανίζουν τα ζώα. Κάποιοι τέτοιοι εκτροφείς ε, πρέπει να τύχουν ηλικής μεταχείρισης ε, και ας ε, μην ξεχνάμε και την σημασία, την κλίμακα. Πρώτα θα ασχοληθούμε με την ανθρώπινη υγεία και μετά με την ζωική υγεία. Και υπάρχουν σοβαρότατα θέματα ψυχικής υγείας. Τώρα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας, ε, δίκιο έχετε. Υπάρχει νομοθεσία και πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Σωστή είναι η επιχειρηματολογία σας. Δεν χρειάζεται να σπεύσουμε να ψηφίσουμε νέα νομοθετήματα πριν εφαρμοστούν τα παλιά. Τώρα, ε, θα ήθελα να ακούσω και την εισηγήτρια και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ε, και εγώ έχω μπερδευτεί. έχω την εντύπωση ότι τα δικά μας τα πρότυπα για την ευμερία των ζώων δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη από τον ΠΟΕ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω. Για το θέμα των αυγών, ε, των παραγωγών ορνήθων και το θέμα των κλοβών, ε, ναι μεν ναι, εξάγονται, ε, μάλλον εξάγεται η παραγωγή, αλλά στην ε, τελευταία θητεία που ψηφίστηκε αυτή η απαγόρευση επειδή ήθελαν την λαϊκή υποστήριξη και π.χ. στους ίδιους εφημερίδες δεν σκέφτηκαν τις επιπτώσεις. Ήταν, πάρα πολύ, ήταν κάκιστη η ιδέα ε, για τους κλοβούς ε, γιατί δεν λάβαμε υπόψη συνέπειες ότι δηλαδή πρόκειτο να εκτοπιστεί η παραγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και ε, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι όλοι είναι υπέρ ε, της ευμερίας των ζώων αλλά δεν θέλω να καθοδηγούμαστε από αυτά τα επιχειρήματα των φιλόζων ε, χωρίς να βασιζόμαστε ε, σε επιστημονικά δεδομένα και να δούμε ε, τι έχει γίνει στον Πούι. Μπορεί να έχει γίνει ένα θαύμα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν νομίζω, αλλά σίγουρα όχι συναισθηματισμοί παρακαλώ. Ο κύριος Κάπλα Σάντος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Είναι σημαντικότητο και πολύ ευαίσθητο αυτό το ζήτημα και πρέπει να το δούμε από δύο διαφορετικές πλευρές. Υπάρχει θέμα πολιτιστικό αφεντός και, αξιών και απ' την άλλη υπάρχει και το οικονομικό ζήτημα. Είναι πολύ καλή η έκθεση, αλλά χωλαίνει γιατί εστιάζεται υπέρμετρα στο δεύτερο σκέλος. Υπάρχει το θέμα της ομότητα, τη ομής συμπεριφορά κατά των ζώων, έτσι, και ακούσαμε διάφορα παραδείγματα. Υπάρχουν κάποιοι που πάσχουν και ε, ε κακοποιούν τα ζώα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και ανάγκη να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή τελικά τι επιβάλλουμε κανόνες που οδηγούν ε, σε χειρότερα αποτελέσματα. Θα ήθελα να μου απαντήσει η συγγήτρια σε δύο ερωτήματα. Ε, ξέρω δεν έχουμε και πάρα πολύ ε, χρόνο, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις, αλλά τέλος πάντων, αν μπορεί να μου απαντήσει για το εξής. Ε, ε, μιλάμε για ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Προστασίας των Η Συνάδελφος το είπε, μέσα στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συγγήτρια ε, ενθαρρύνει την δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ποια θα είναι τα καθήκοντά του. Ούτε στην έκθεση τη ηγήτρια, ούτε στο έγγραφο ανατολισμό τη Επιτροπή ε, διευκρινίζεται ακριβώ ποια θα είναι τα καθήκοντα αυτού του Ευρωπαϊκού ε, Κέντρου. Ε, Μήπω ε, απορροφήσει κονδύλια χωρί να ξέρουμε ποιε υπηρεσίε θα παράσχει ή η συγγήτρια ή η η Επιτροπή. Παρακαλώ να μου εξηγήσουν ακριβώ τι θα κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την προστασία των ζώνων. Ευχαριστώ, Λουί. Ο Μάρτιν τώρα. Ναι. Ναι, κυρία Πάλσουν, και εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Συμφωνούμε σε πολλά σημεία μαζί σα. Θα ήθελα απλώ να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Από τη μία υποστηρίζουμε ρητά τη στάση σα ότι χρειαζόμαστε ίδιες προδιαγραφέ σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη ε, χρειαζόμαστε ένα επαρκέ σύστημα ελέγχου. Ε, συμφωνούμε πολύ μαζί σα. Δεν είναι δυνατόν προ τα έξω να ζητούμε προστασία και να μην τηρούμε εντό τη Ευρώπη τι ίδιε μα τι προδιαγραφέ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά το μέλλον. Θα ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ με πολλού συναδέλφου που θεωρούν ότι η προστασία των ζώων επιβαρύνει τη γεωργία. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το έμβλημα τη Ευρωπαϊκή Γεωργία ότι φροντίζει για την ευημερία των ζώων. Ε, δικαιολογημένα θίξατε το ζήτημα των αντιβιωτικών ε, και το θέσατε στο επίκεντρο τη συζήτηση αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε τόσο θαραλέοι για να συζητήσουμε για την συγκέντρωση στον τομέα της προστασίας των ζώων. Εκεί που είναι οι οι συνθήκες εξασφαλίζεται η ευημερία των ζώων. Αλλά εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη πυκνότητα όπως ισχύει για τις όρνηθες αλλά και για τους ε, ε, χείρους ε, εκεί αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε προβλήματα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ε, προβλήματα δηλαδή που αφορούν τη μαζική εκτροφή των ζώων. Και όταν μιλούμε για αντιβιωτικά θα πρέπει να μιλήσουμε για τα αντιβιωτικά σε σχέση ακριβώς με αυτό το φαινόμενο μαζικής εκτροφής ε, ζώων. Νομίζω ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση συνδέοντας δηλαδή τα δύο ζητήματα. Äh, Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πάλσεν για την έκθεσή της. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα ήθελα απλώ να συμπληρώσω κάτι. Κατά, σύμφωνα με την εμπειρία μου, όταν θέλουμε να κερδίσουμε τον Γεωργό σαν σύμμαχο όσον αφορά την προστασία των ζώων, ε, Ε, τι συμβαίνει όταν τον... Ε, ε, μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά τον εξοργίζουμε τον Γεωργό όταν βλέπει ότι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν, άλλοι, υπάρχουν άλλες προδιαγραφές. Και μετά έχουμε εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματικά δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις προδιαγραφές. Αυτό εξοργίζει τους Γιωργούς. Ε, και κάτι άλλο, χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω η προστασία των ζώων, αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτε σε αυτό το οποίο απαιτούμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζεται και για τι εισαγωγέ. Αυτό συνδέεται και με την προστασία των καταναλωτών. Γιατί ο καταναλωτή έχει το δικαίωμα όταν αγοράζει ένα προϊόν να γνωρίζει ότι το ζώο από το οποίο προέρχεται το προϊόν έχει εκτραφεί με τον σωστό τρόπο. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να πούμε ε, λίγα ζώα εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό προστασίας ή η μαζική εκτροφή ε, δεν μπορεί να συνοδεύεται από σωστή προστασία των ζώων. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όσον αφορά τα αντιβιωτικά, Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη μεμονωμένα για το κάθε ζώο. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να εξοραίζουμε τα πράγματα γιατί αυτό μας οδηγεί σε μια εσφαλμένη κατεύθυνση. Λοιπόν, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνατότητα ελέγχου των διατάξεων, της εφαρμογής των διατάξεων και προστασία, υψηλό επίπεδο προστασίας και στις ε, τρίτες χώρες. Αυτά τα τέσσερα σημεία νομίζω ότι θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόπιτς τώρα. Ο Ντόν Ρούμπιξ. Έχω να κάνω διάφορα σχόλια. Φυσικά είμαι υπέρ της ευημερίας των ζώων Πρέπει να αφαιρόμαστε ανθρώπινα ε, στα ζώα που μας ε, προσφέρουν ε, την τροφή που καταναλώνουμε. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στα ζώα και πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τις ζωικές τροφές Παραδείγματο χάρη, έχουμε μετατρέψει την Αγελάδα σε γαλακτοπαραγωγική μηχανή και στη συνέχεια τη φάζουμε κιόλα για κρεατοπαραγωγή. Αλλά οι αγελάδες αυτές δεν μπορούν να είναι στα λιβάδια ελεύθερες, τους δίνουμε να φάνε οτιδήποτε, μετά τις πετάμε μέσα σε φορτηγά, τις αρμέγουμε και τις φάζουμε κιόλας. Στη Λετωνία, εσχάτως, ε, έγινε μία μελέτη βάσει της οποίας ε, γενετικά τροποποιημένα φασόλια χρησιμοποιούνταν για, ως ζωοτροφές και φυσικά περάσανε κάποια στοιχεία γενετικώς τροποποιημένα ε, στο γάλα και ε, αντίστοιχα πέρασαν αυτά τα στοιχεία ε, στις γυναίκες, σε γαλοχούσες γυναίκες που στη συνέχεια νόσησαν. Εσείς μιλήσατε για πάνθρωπους ε, αστα... Ε, ψυχικά και πνευματικά ασταθείς ανθρώπους που κακοποιούν τα ζώα. Δηλαδή εμείς είμαστε καλύτεροι με αυτά που δίνουμε στις αγελάδες ε, να φάνε. Ενώ ξέρουμε ότι μεταδίδονται νόσοι. Νομίζω πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε κατά νου εξετάζοντας τη συγκεκριμένη έκθεση. Vă mulțumesc. Doamna Calniete, aveți Καλνίεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίως να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές, στην εισηγήτρια μάλλον, γιατί νομίζω ότι η έκθεση αυτή μας δείχνει το τι ακριβώς έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης το οποίο έχει γίνει δεκτό. Έχει μεγάλη σημασία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά με, ε, με ομοιογενή τρόπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό θα ήταν το σύστημα αυτό να ίσχυε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά Εν πάση περιπτώσει είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Πάντως δεν χρειαζόμαστε μια καινούργια υπηρεσία για να επιδιώξουμε κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Σχετικά με τη νέα υπηρεσία θα ήθελα να μάθω πόσο θα κοστίσει στους φορολογούμενους, τι λειτουργίες θα έχει και τι δικαιώματα θα έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία την οποία προτείνεται να δημιουργηθεί. Όπως και προηγούμενοι ομιλητές θα ήθελα να πω ότι έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση η παραγωγή, η κτηνοτροφία γενικότερα, ιδιαίτερα σε σχέση και με το τι κάνουν τρίτες χώρες, οι οποίες θα πρέπει να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά διασφάλισης ποιότητας γιατί αλλιώς οι γεωργοί μας δεν θα είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστικοί όπως η γεωργοί από άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν γενικά γεωργοί οι οποίοι παράγουν γεωργικά προϊόντα χωρίς να υπακούν σε τέτοιου είδους, ε, ε, σε τέτοιου είδους κανόνες και νόμους όπως η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοώ την ευθύνη την οποία δείχνουν οι συνάδελφοι σχετικά με την ένταξη και των οικιακών, των κατοικιδίων συγγνώμη Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Τώρα μιλάμε για τα βοηδή, τα πουλερικά, τους χείρους. Αυτά είναι τα ζώα τα οποία σε αυτή τη φάση μας απασχολούν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε δυσκολότερη τη ζωή ε, των ανθρώπων που έχουν ε, τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες. Δεν θέλουμε εμείς να παρέμβουμε σε θέματα που αφορούν τα κατοικίδια. Ευχαριστώ πολύ. έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο κόσμος να μάθει να πεπατά πριν αρχίσει να τρέχει. Ας δούμε κάποιες από τις κοινοτικέ προτάσεις. Η μία αφορά τη μεταφορά των ζώων. Εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω τα πρόβατά μου ε, περισσότερο από 33 ε, μίλια μακρύτερα από το, από το κτήμα μου. Η γυναίκα μου έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, μπορεί να ελέγχεται, έχει περάσει το τεστ, αλλά αν τη σταματήσει η αστυνομία και έχει ξεπεράσει τα μίλια τα οποία δικαιούται να κάνει μεταφέροντα ζώα θα διωχθεί ποινικά. Όταν τα λέω αυτά σε άλλους φίλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κοιτάνε περίεργα, μου λένε μα είστε τρελοί εσείς που κάνετε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν τέτοιου είδους κανόνες εφόσον τους επιθυμούν να τους εξηγήσουν και να ισχύσουν για όλους. Τα προβλήματα θα ξεκινήσουν για τα πουλερικά σε 8-9 μήνες όταν θα γεννηθούν τα νέα μικρά κοτόπουλα. Κανονικά θα πρέπει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάψουν να παράγουν αυγά από οτό και σόρνηθες σε συστοιχίες κλοβών. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα συνεχίσουν να το κάνουν παρά το ότι κάποιοι από τις παραγωγείς τους πήραν επιδοτήσεις κατά 50% για να αλλάξουν τα συστήματα παραγωγής που δεν ισχύει για μας. Και μετά το 2012 οι παραγωγοί σε αυτές τις χώρες μπορούν να πολλούν τα ΟΑ στους καταναλωτές στη Μεγάλη Βρετανία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό πραγματικά θα μειώσει την εμπιστοσύνη προς τον Βρετανό παραγωγό και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τους επιβαρύνουμε με περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να βοηθήσουμε πράγματι, γιατί όπως είπε ο Ιρλανδός συνάδελφος, όταν συμβεί αυτό που περιμένουμε το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι έτοιμη. Η παραγωγή αυγών στην Ιταλία και την Ισπανία δεν θα μπορέσουν ε, να αλλάξουν και θα υπάρξει έλλειψη γιατί οι καταναλωτές θα θέλουν πάντα τα ίδια αυγά να καταναλώνουν. Από πού θα τα εισάγουμε, από την Ινδία, από την Ουκρανία και αυτά τα αυγά θα προέρχονται από τόκες όρνηθες σε κλωβούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει τεράστιες δαπάνες και προσπάθειες για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά για να πείσουμε τους καταναλωτές να μην προτιμούν τα εισαγόμενα προϊόντα. Ευχαριστώ. Να σας διαβεβαιώσω αγαπητές συνάδελφοι ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία ήδη είναι απόλυτα συμβατές με τους κοινοτικούς ε, ε, νόμους και ρυθμίσεις. Η μεταβατική περίοδος την οποία αναφερθήκατε ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της ένταξης ε, των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω το λόγο στον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πάλσεν για την εργασία της. Αλλά ήθελα να πάρω το λόγο κυρία Πάλσεν γιατί στην αρχή της ομιλίας σας είπατε ότι έχω βαρεθεί να βλέπω αυτές τις ε, ταινίες όπου παρουσιάζονται οι παραβιάσεις κατά των ζώων. Εγώ γνωρίζω μια ταινία η οποία προβάλλεται εδώ και 30 χρόνια. Στη γερμανική τηλεόραση προβάλλεται αυτή η ταινία. Υπάρχει μια, ε, ένα πλοίο με μια αγελάδα που είναι κρεμασμένη από τα πόδια και η ταινία αυτή προβάλλεται ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε με αυστηρέ διατάξει για την προστασία των ζώων, αλλά ακόμα και οι πιο αυστηρέ διατάξει δεν μπορούν να εμποδίσουν τι ε, παραβιάσει θα, πρέπει να, ε, θα υπάρχουν και στο μέλλον μεμονωμένες περιπτώσεις όπου θα σημειώνονται αυτές οι παραβιάσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και ήθελα να πάρω το λόγο γιατί ο κύριος ε, Χόισλινγκ ε, μίλησε για τη μαζική εκτροφή των ζώων. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτές τις διατυπώσεις. Ε, μπορεί κανείς να κακομεταχειρίζεται και μία αγελάδα και να φέρετε πολύ καλά σε 400 αγελάδες. Ο πατέρας μου ήταν ε, και μελισσοκόμος. Ε, και ε, στις, οι μέλισσες ε, ε, ζουν μαζικά. Υπάρχουν τεράστιοι αριθμοί μελισσών. Άρα λοιπόν η ίδια η φύση μπορεί να εξασφαλίσει παρά τους υψηλούς αριθμούς στον πληθυσμό των ζώων σωστές ε, προδιαγραφές ευημερία. Τώρα, όσον αφορά τις επραγματεύσεις με τον ΠΟΕ, γίνονται σχετικά πολλές συζητήσεις, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΟΕ δεν έχει σοβαρή πρόθεση να συμπεριλάβει το θέμα στην ημερήσια διάταξή του. Ε, και νομίζω θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση ε, και στην Επιτροπή Ίντε, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό και να έχει την προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις. Ο Στεφάν Λεφόλ έχει το λόγο. Ναι, θα είμαι ε, σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η βάναυση μεταχείριση των ε, ζώων υπάρχει, αλλά καμιά φορά οι άνθρωποι είναι βάναυση και με τους ίδιους αυτούς τους. Και ε, δεν θα πρέπει να το λησμονούμε, γιατί έγιναν εδώ κάποιες παρατηρήσεις που λένε ότι αυτή η συζήτηση για την ευημερία των ζώων ε, θα πρέπει να βασίσετε σε μια αντίληψη του ανθρωπισμού. Ε, ο ανθρωπισμό θα πρέπει να ισχύει για τα ζώα και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Λοιπόν, εάν χρειαζόμαστε μια εναρμόνιση των κανόνων και εγώ είμαι υπέρ, θα ήθελα όλοι όσοι διεκδικούν κάτι τέτοιο σήμερα να έχουν τι ίδιε ανησυχίε όταν μιλούμε, για παράδειγμα, για κοινωνικά θέματα, για τι κοινωνικέ πτυχέ. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια χώρα. Όσον αφορά τι ε, προτάσει που έκανε η κυρία Πόλσον και θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο Λουί Καπούλα Σάντο για το στόχο ενό παρατηρητηρίου, για του στόχου, συγγνώμη, ενό παρατηρητηρίου παρατηρητηρίου. Για παράδειγμα, τον καθαρισμό κανόνων και το ρόλο της Επιτροπής. Δεν θα είναι ένα παρατηρητήριο το οποίο θα βρει κάποιες λύσεις. Στο επίπεδο των ε, κανόνων, εδώ γίνεται η συζήτηση. Ε, σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να γίνει η εναρμόνιση και εδώ θα πρέπει να είναι όλοι σύμφωνοι. Το επίπεδο όπου κανένας μπορεί να εκφράσει μία άποψη για την ευημερία των ζώων θα καθορίσει και το επίπεδο εναρμόνισης ευρωπαϊκή κλίμακα. Ε, τώρα, όσον αφορά το ΜΠΟΕ, όταν μιλάμε για την ευημερία των ζώων και δεν μπορούμε να συζητήσουμε ούτε για τις κοινωνικές προϋποθέσεις ε, ούτε για τις περιβαλλοντικές προϋπεθέσεις και λέμε ότι θα διαπραγματευτούμε παρόλα αυτά με τον ΠΟΕ, νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τους ε, εαυτούς μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την διαχείριση του κόσμου. Εγώ είμαι υπέρ της ευημερίας των ζώνων, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε νυφάλοι και διαβίσεις όσον αφορά ε, τον ΠΟΕ και θα πρέπει η βούληση εναρμόνιση των κανόνων να τεθεί στο επίπεδο ή στο ύψος όπου η κάθε χώρα προσλαμβάνει τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και ζώου και ακριβώς με τον τρόπο που ορίζει αυτή τη σχέση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την εργασία της κυρίας Πούλσον. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Αξιολόγηση του προγράμματος δράσης 2006-2010». Αυτό το κομμάτι το βρήκα σχετικά συνοπτικό συγγνώμη, στην έκθεση αυτή. Αναλύει βέβαια τα κείμενα τα οποία παρήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά θα ήθελα μια πραγματική αξιολόγηση του τι συμβαίνει, να δούμε ποιες είναι πραγματικά οι δυσκολίες, γιατί δεν έχουμε προχωρήσει με το ρυθμό τον οποίο θα έπρεπε στο σύνολο της Ένωσης και τι πρέπει να διορθώσουμε για να εφαρμοστεί η σημερινή νομοθεσία πριν φανταστεί κανείς νέα στάδια νομοθετικά, αν είναι απαραίτητα. Γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο για πάρα πολύ κόσμο. Διάβασα βέβαια την έκθεση αυτή όταν είδα τις πρώτες εικόνες από την ΑΕΤ και αυτό με ενόχλησε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ κύριε Νταντέ. Τέλειωσε η συζήτηση και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Πόλσον. Τελικές παρατηρήσεις κυρία Πόλσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Ήλπιζα ότι θα συζητούσαμε την, το ζήτημα της προστασίας και της ευημερία των ζώων αυτό καθε αυτό. Νόμιζα ότι υπήρχε συνένεση ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε τη λογική μεταχείριση των ζώων και την αξιοπρεπία στη μεταχείρισή τους. Και το θέμα μας ήταν στην πράξη τι θα γίνει. Πώς ακριβώς μπορούμε να έχουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού πρώτα απ' όλα στην ενδοκινοτική αγορά. Πώς ακριβώς θα τα καταφέρουμε με τις οικονομικές προκλήσεις. Πώς ακριβώς ε, θα εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ε, και την συμμόρφωση με τις αποφάσεις που έχουμε λάβει. Για μένα είναι πρακτικό το ζήτημα εφαρμογής από την κοινωνία της νομοθεσίας. Είναι τόσο λίγοι αυτοί οι εκτροφείς που κακοποιούν τα ζώα. Εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει κανέναν. Υπάρχουν μικρές μονάδες όπου οι εκτροφείς φροντίζουν τα ζώα. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλες μονάδες ε, καταδεικνύουν ότι εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή διαβίωση στα ζώα. Νομίζω ότι συμφωνούμε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με τον υπόλοιπο κόσμο εάν δεν ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις. Μετά περνάμε στα τεχνικά ζητήματα. Δεν θέλω, δεν επιθυμώ εγώ την ίδρυση νέου φορέα. Εγώ μιλώ για τον έλεγχο. Ο ΦΑΟ, παραδείγματο χάρη, έχει επαρκεί πόρου. Έχουμε τον ΕΦΣΑ που ρυθμίζει ζητήματα όπως η αντοχή στα αντιβιωτικά. Δεν προτείνω εγώ την ίδρυση νέας αρχής για την τεχνική ανάπτυξη, για την έρευνα, για το συντονισμό των επιστημονικών γνώσεων. Ναι, έλεγα ότι ίσως κάποιο εθνικό Ινστιτούτο από κάποιο κράτος μέλος ή μία υπηρεσία της Επιτροπής μπορεί να αναλάβει αυτό το έργο δεν ε, διανοούμε εγώ ίδρυση νέου φορέα αν δεν συντονίσουμε πρώτα τη δράση των υφιστάμενων οργανισμών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλό είναι που μπορέσαμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Ευχαριστώ την κυρία Πόλσον για την εξαιρετική προσπάθεια. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε αργότερα στη συζήτηση αυτή. Κλείνω το, τη συζήτηση θυμίζοντας ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 12η Μεσημβρινή. Περνάμε τώρα γρήγορα στην τελευταία ε, έκθεση την οποία έχουμε για σήμερα. Το θέμα της καλύτερης ε, λειτουργίας ε, της αλυσίδας των τροφίμων στην Ευρώπη είναι μια πρώτη συζήτηση την οποία κάνουμε σήμερα. Θα ζητήσω από τον εισηγητή, τον Ζωζέ Μποβέ, να κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα. Είδαμε ότι πολλές φορές οι διακυμάνσεις των τιμών δημιουργούν πολλά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο βέβαια για να μπούμε στην ουσία που θα επιθυμούσαμε και γι' αυτό ζητώ από τον κύριο Μποβέ να κάνει μια συνοπτική παρουσίαση και να ακούσουμε μετά τις απόψεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφόσον το επιθυμούν. Ζωζέ Μποβέ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κοιτάξτε τώρα ναι, άμα έχουμε μόνο λίγα λεπτά θα δυσκολευτούμε. Πώς θα γίνει η συζήτηση. Να ακούσουμε και τους εκπροσώπους Επιτροπής. Για μένα το σημαντικό είναι να εμπλουτίσουμε τις προτάσεις μας και τα επιμέρους, ε, κεφάλαια, τα επιμέρους ζητήματα μάλλον θέλουμε να προωθήσουμε δια τις συζητήσει που θα κάνουμε. Αν τώρα δεν γίνεται να το συζητήσουμε το θέμα, επειδή είναι σχεδόν έξι και έχουμε την συνεδρίαση στη συνέχεια, το αφήνω στα χέρια σας. Μήπως να το αναβάλουμε για αύριο, μήπως για την επόμενη συνεδρίαση, για να κάνουμε ταυτόχρονα την παρουσίαση, τη συζήτηση με την Επιτροπή και τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Παρά είναι σοβαρό το ζήτημα για να το περάσουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την άποψη. Πράγματι για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ευχαριστώ τον Ζωζέ Μποβέ. Λοιπόν θα το συζητήσουμε σε μια επόμενη συνεδρίαση. Τώρα θα πρέπει να κλείσουμε την σημερινή συνεδρίαση. Θυμίζω ότι αύριο φιλοξενούμε την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, την κυρία Ελένη Εσπινόζα. Και αύριο η συζήτησή μας θα ασχοληθεί με τα θέματα των κλιματολογικών αλλαγών. Οι συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα, συνεχίζουν τη συνεδρίαση